Good afternoon to uh, everybody. Καλησπέρα σε όλους. Ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το τελευταίο κομμάτι της ε, συνεδρίασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών που είναι διήμερη και βέβαια καλωσορίζω θερμά τον Υπουργό ΟΓΟΤ τον οποίο και ευχαριστώ θερμά που δέχτηκε την πρόσκλησή μας ε, σήμερα εδώ. Θεωρώ πως ε, πρόκειται για μια συζήτηση που γίνεται στην κατάλληλη χρονική συγκυρία, γιατί η γερμανική διαπραγμάτευση ξεκίνησε ε, την περασμένη εβδομάδα σε ό,τι αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ο χρόνος μας πιέζει και η προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει στο μέλλον της αλλά και να υποστηρίξει και μια ανάκαμψη η οποία θα είναι και βιώσιμη και ανθεκτική. Να υπενθυμίσω ε, εδώ ότι το Κοινοβούλιο από την Πράτου ξεκίνησε αυτή τη διαπραγμάτευση με διαλλακτικό πνεύμα ε, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Ε, αναμένουμε βέβαια περισσότερα σε ό,τι αφορά το κομμάτι δικότερα των εσόδων, αλλά θα δείξουμε καλή θέληση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το να περάσει γρήγορα η δική μα γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά την απόφαση για του ιδίου πόρου, έτσι ώστε να υπάρξει και η δική μας γνώμη συγγνώμη σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους και τη σχετική απόφαση έτσι ώστε να περάσουμε σε ταχεία εφαρμογή της, ε, του σχεδίου ανάκαμψης. Και γι' αυτό αναμένουμε από δική σας πλευρά κύριε Υπουργέ μια ανοιχτή στάση έτσι ώστε να διευκολύνουμε την πολιτική συμφωνία και τελικά να δώσει τη συμφωνία του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη συνενέση του. Εάν τελικά δεν εμ, πληρωθούν τα δικά μας αιτήματα έως τα τέλη Οκτωβρίου θα ε, προχωρήσουμε στο σχέδιο ε, έκτακτη ανάγκη μα, αν θέλετε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα συμφωνήσουμε επί του προπολογισμού του 2021 ε, και επί των προγραμμάτων του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου σε, με βάση ε, τα ανώτατα όρια του 2020, όπως αυτά θα επιταθούν για το 2021 και τις τρέχουσες διατάξεις του τρέχοντος δηλαδή του ισχύου του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά από την πλευρά μου κύριε Υπουργέ και έχετε τώρα το λόγο για να κάνετε τα δικά σας σχολεία για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ε, θα ήθελα και εγώ βέβαια να βρίσκομαι σήμερα ε, ε, στις Βρυξέλλες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα έτσι όπως έχουν και κατάσταση με την πανδημία δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ και με τη φυσική δηλαδή μου παρουσία σε μια συνεδρίαση μαζί σας. Για, μας, για μένα συγκεκριμένα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και με τη δική σας Επιτροπή, την Επιτροπή Προϋπολογισμών, γιατί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και το όλο πακέτο για την ανάκαμψη αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο για την ανάκαμψη των κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης ε, με ενδιαφέρει ε, πολύ να αναδείξω εδώ τον αποφασιστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ ε, και 22 χρόνια εγώ είμαι ε, βουλευτής ε, και θεωρώ πραγματικά πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα εταίρο μας, ένα ισχυρό εταίρο και όχι αντίπαλο μας. Καθώς είχα ήδη σήμερα τη δυνατότητα να συζητήσω με ε, μέλη άλλη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να το τονίσω αυτό για μία ακόμα φορά. Ότι δηλαδή εδώ δεν τοποθετούμε εκ μέρου ε, τη γερμανική κυβέρνηση και δεν εκπροσωπώ εδώ κάποια πολιτική ομάδα ή κάτι άλλο. Όχι. Μιλώ μαζί σα σήμερα εδώ με την ιδιότητα του προσώπου του Συμβουλίου. Άρα λοιπόν τα όσα θα σας πω ε, αποτελούν άποψη 27 κρατών μελών κρατών μελών τα οποία ε, εκπροσωπούνται ακριβώς ε, μέσω του Συμβουλίου, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε εύκολο. Και επίσης ε, με χαροποιεί το γεγονό ότι υπάρχουν μεγάλε και υψηλέ προσδοκίε σε ό,τι αφορά την Προεδρία τη ε, Γερμανία στο Συμβούλιο. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι υπάρχει και μεγάλη εμπιστοσύνη απέναντί μα. Και ε, στο πλαίσιο των συνομιλιών που είχα με διάφορου ευρωβουλευτέ, διαπίστωσα ότι υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη, αυτή η βάση εμπιστοσύνη και ε, ελπίζω να συμβάλλω και με την συζήτηση σήμερα εδώ σε αυτή την εμπιστοσύνη έτσι ώστε να διασφαλίσουμε και την απαραίτητη σταθερότητα για την επόμενη φάση. Και αυτή η σταθερότητα είναι απαραίτητη γιατί όπως το ανέφερε μόλις ε, τώρα και ο Πρόεδρος, οι διαπραγματεύσει που μας περιμένουν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Με την πανδημία του COVID έχουμε να κάνουμε με μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις ε, στην ιστορία της ΕΕ. Ταυτόχρονα έχουμε μία, ένα πολυπολικό αν θέλετε κόσμο, μία πολυπολική ε, τάξη πραγμάτων, η οποία μάλιστα δέχεται μεγάλες πιέσεις και επίσης από εκεί και μετά η δική μας γενιά ε, έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει τις ε, προϋποθέσεις και τις συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ανάκαμψη ε, του, του κλίματος, δηλαδή για την, τη λήψη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος και από εκεί και μετά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να αναλάβει το ρόλο ε, που τη αντιστοιχεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μια ε, οικονομική νομισματική ένωση, δεν αποτελεί μια κοινή αγορά. Ε, αποτελεί μια ένωση αξιών και αρχών. Τώρα, η δέσμη την οποία συζητούμε σήμερα εδώ, η δέσμη προτάσεων, το πακέτο αυτό, σίγουρα ε, συμφωνήθηκε ε, στο πλαίσιο ε, πολύ μεγάλων δυσκολιών και πιέσεων που ασκήθηκαν. Όπως γνωρίζετε, αποτέλεσε το αποτέλεσμα μιας ε, συνεδρίασης που ήταν από τις δυσκολότερες και από τις πιο... Ε, από εκείνες που διήρκεσαν περισσότερο στην ιστορία του Συμβουλίου. Υπήρξαν διαφορετικές τοποθετήσεις, χάσμα μεταξύ διαφορετικών απόψεων, υπάρξαν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα και δείξαμε με αυτόν τον τρόπο και δώσαμε το στίγμα της αλληλεγγύης μας. Και πραγματικά για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα χρειάστηκε όλοι να δείξουν διαλλακτική στάση και όλοι να προβούν σε κάποιους συμβιβασμούς. Ε, νιώτε ε, επίπονος. Όμως χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη όλων για όλα τα κομμάτια. Δηλαδή σημαίνει ότι το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα και το Next Generation EU αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία θα πρέπει να ιδωθούν ως ένα κοινό πακέτο. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε επιμέρους στοιχεία ξεχωριστά το καθένα. Ε, θεωρώ δηλαδή πως κάτι τέτοιο θα ε, καθιστούσε ουσιαστικά αδύνατη διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο. Θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού ως δέσμη όλα αυτά τα Όλε αυτές τις προτάσεις. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω εμφατικά εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ε, δώσατε την απαραίτητη όθηση σε αυτή τη διαδικασία, θέσατε πολύ σημαντικά ζητήματα για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση, των, ε, την αύξηση δηλαδή των κοντιλίων σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή αλλά ταυτόχρονα δώσατε πολύ μεγάλη έμφαση στα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα πράγμα το οποίο μερικές φορές ήταν δύσκολο να το κάνουμε στις διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο. Πάντω, σημαντικό σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του αποτελέσματο που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μα είναι το ότι το να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτός ο συμβιβασμό ε, δεν θα πρέπει να ε, αξιολογηθεί ακριβώς με βάση ε, τις αξιώσεις που είχαν τεθεί πριν από κάποια χρόνια υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Νομίζω πως το αποτέλεσμα από μόνο του καταδεικνύει την αξία του και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα επιμέρους στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά όχι μόνο για μας το Συμβούλιο αλλά και για σας νομίζω ως Κοινοβούλιο. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό αυτού του, αυτού του συμβιβασμού ε, στο μέλλον. Ναι, υπήρξαν κάποιες κριτικές, αλλά για παράδειγμα, τα ε, κονδύλια για το Erasmus Plus, ένα πρόγραμμα εξαιρετικά σημαντικό για όλους μας, αυξάνονται κατά 50%. Σε ό,τι αφορά το Horizon ε, Europe, έχουμε αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά σχεδόν 25%. Ταυτόχρονα ενισχύουμε τις πράσινες και ψηφιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους, έχουμε επιτύχει, έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ε, βρισκόμαστε σε μια καμπή νομίζω εδώ. Έχουμε καταρχήν ε, την επιβολή του φόρου για τα πλαστικά από το 2021, δημιουργώντας ακριβώς ένα νέο είδος ιδιοπόρου αν θέλετε, το οποίο θα ε, θα έρθουν να συμπληρωθούν και κάποια ακόμα και από εκεί και μετά κάτι εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός το ότι ε, το 30% των κοντιλίων θα ε, δεσμευθεί για τους στόχους της ε, κλιματικής αλλαγής. Δεν υπάρχει νομίζω εθνικός προϋπολογισμός ο οποίος να είναι διαρθρωμένος με αυτόν τον τρόπο, να δίνει δηλαδή τόση σημασία στην κλιματική αλλαγή. Από εκεί και μετά ένα ακόμα πολύ σημαντικό και για το Συμβούλιο ζήτημα είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Ποιο θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό που επιτύχαμε, ότι δηλαδή επιτύχαμε ακριβώ μια τέτοια προπόθεση, μια αίρεσιμότητα σε ό,τι αφορά ε, την, ε, την επιβολή του κράτου δικαίου, προκειμένου να προστατεύσουμε και το προπολογισμό μα. Αποτελεί κάτι τέτοιο νομίζω επιτυχία, αλλά αποτελεί και καμπή ε, για μα. Και ενδεχομένω ναι, υπάρχουν και κάποια περιθώρια σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των όσων συμφωνήθηκαν, αλλά νομίζω πω έχουμε ξεκινήσει σωστά και νομίζω πως σε τέσσερις εδώ πολιτικές ομάδες ε, του Κοινοβουλίου τόνισαν το, ε, τη σημασία ε, που έχει για αυτές, αυτή η αιρεσιμότητα, αυτή η προϋπόθεση σε ό,τι αφορά την κρίση του κράτους δικαίου. Παρ' όλα αυτά, το Συμβούλιο τώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να φτάσουν σε μια συμφωνία σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη εφαρμογή στην πράξη του σχετικού κανονισμού. Και γι' αυτό θα χρειαστεί και η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και το σύνολο των κρατών μελών από την πλευρά του Συμβουλίου. Πράγμα το οποίο δεν θα είναι τόσο εύκολο. Οπότε, ε, πραγματικά στο τέλο, ε, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία θα είναι φιλόδοξη, αλλά τελικά που θα είναι και μια λύση με την οποία, την οποία θα μπορέσουν να αποδεχτούν όλοι. Και ε, νομίζω πω και ο πρόεδρος Αλμισελ εδώ ήταν διαθέσιμος απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για περαιτέρω συζητήσεις ε, μαζί σας, αλλά ε, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι από την πλευρά του Συμβουλίου που θα είναι στη διάθεσή σα για περαιτέρω διαπραγμάτευση και εγώ από την πλευρά μου δεσμεύομαι ότι θα είμαι στη διάθεσή σα για περαιτέρω συζητήσει. Εκείνο πάντως που χρειαζόμαστε κυρίε και κύριοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή είναι μια ταχεία ε, συμφωνία σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό γιατί. Γιατί υποσχεθήκαμε στους πολίτες μας ότι τα απαραίτητα μέτρα ε, για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ε, πανδημίας αλλά και τις οικονομικές θα να τεθούν το ταχύτερο δυνατό. Χρειαζόμαστε λοιπόν τι απαραίτητε επενδύσει στην έρευνα, στην υγεία και στι υποδομέ. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στι φιλοδοξίε μα στο επίπεδο τη κλιματική αλλαγή ε, και τη ψηφιακή ε, μετάβαση. Και για αυτόν τον λόγο, ε, κατά την υπόλοιπη διαδικασία τώρα και τα επιμέρου διαδικαστικά στάδια, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο εξή σε ό,τι αφορά τη συμφωνία για του ίδιου πόρου, η οποία θα χρειαστεί να λάβει και την υποστήριξη από πλευρά των κρατών μελών, χρειάζεται χρόνο. Ε, ε, δεν πρόκειται δηλαδή για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσαμε να διευθετήσουμε μέσα σε ε, μέρες ή εβδομάδες. Θα χρειαστούν μήνες και σας το λέω αυτό και με βάση την εμπειρία που έχω και εγώ ως ε, βουλευτής στο δικό μου Εθνικό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, που θα χρειαστεί συμφωνία μεταξύ της Άνω και Κάτω Βουλής. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος και γι' αυτό η προσέγγιση που εμείς ακολουθούμε είναι να εξετάζουμε ως πακέτο το πολιτικές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και ε, τους ίδιους πόρους και από την άλλη πλευρά να λέμε ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχουμε ως στόχο το να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Αλλά και οι διαπραγματεύσει για τι τομεακέ ε, πράξει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με το τέλο του χρόνου. Για άλλη μια φορά, αυτό που θέλω να ζητήσω από εσά είναι, επειδή είμαστε πρόθυμοι νύχτα μέρα να ε, συνεργαστούμε και να διαπραγματευτούμε, να επιδιώξουμε από κοινό μια καλή λύση. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει τώρα είναι να επιτρέψουμε το business as usual. Οι καταστάσεις που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Θα πρέπει λοιπόν ως θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να τις φέρουμε εις πέρας. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη εκεί που χρειάζεται επιγόντως. Ε, γι' αυτό σας ζητώ θερμά υποστηρίξτε μας Δεν σας είπα, δεν ήρθα εδώ όμω να σας πω ε, πώς θέλουν να διαπραγματευτούν οι διαπραγματεύσεις ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Next Generation EU, αλλά οπωσδήποτε είμαι εδώ για να ακούσω και τις δικές σας απόψεις και τοποθετήσεις και να δούμε πώς από τις διαπραγματεύσεις θα φτάσουμε σε ένα κοινό αποτέλεσμα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Υπουργέ Ροτ για αυτές τις ε, εισαγωγικές παρατηρήσεις ό,τι αφορά τη διοργάνωση της συζήτησή μας. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε ε, τους, ε, τα μέλη της δημοτευτικής ομάδας, τρία λεπτά ο καθένας, και μετά τους κοιόδης εισηγητές. Και στο βαθμό που θα επιτρέψει ο χρόνος, γιατί στις 6 θα σταματήσει η διερμηνία, θα έχουμε και τις παρεμβάσεις των υπολείπων μελών. Για τη διαπραγματευτική λοιπόν ομάδα, πρώτα απ' όλα ο κύριος Όλμπριχτ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, για την ε, δυνατότητα που μας δίνεται να αλλάξουμε απόψεις. Όπως γνωρίζετε, μετά την πρώτη συνάντηση, ε, όχι τριλόγο αλλά τριμερούς διαλόγου, όπως είπε και ο πρέσβης, ε, αναμένουμε τις επόμενες συναντήσεις και μπορούμε να πούμε, νομίζω αυτή τη στιγμή, ότι συμμεριζόμαστε πολλά από αυτά που αναφέρατε. Δηλαδή και εμείς θέλουμε τα πράγματα να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ε, η προσέγγιση μας είναι κοινή, διότι όλοι περιμένουν αποτελέσματα, περιμένουν σαφήνεια. Ταυτόχρονα, αυτό το λέγαμε και πριν τις διαπραγματεύσεις, ε, αλλά οι διαπραγματεύσεις πρέπει να οδηγήσουν ε, σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποιους συμβιβασμούς. Τα συμπεράσματα όμως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μπορεί να είναι μια κάποια εντολή για τους υπουργούς ε, για την διαπραγμάτευση. Εμείς έχουμε όμως το δική μας εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ψήφισμά του. Νομίζω λοιπόν ότι και οι δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσουν με βάση την εντολή που έχουν λάβει. Βεβαίως ε, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν εξαιρετικά σημαντική ε, και ήταν εξαιρετικά σημαντική για να αλλάξει όλη η δομή ε, του συστήματος ε, του δημοσιονομικού για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση. Όμως, όπως ξέρετε και εσείς και εμείς, αυτό το πακέτο είναι το MFF PDP ε, συν το σχέδιο ανάκρισης, συν κράτος δικαίου. Εφόσον αυτό είναι το πακέτο, θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς συνδέονται μεταξύ τους τα διάφορα στοιχεία αυτού του πακέτου. Μπορούμε να δεχτούμε δηλαδή ένα μέρος του πακέτου και μετά το άλλο και μετά το τρίτο. Το πραγματικό ερώτημα είναι, παραδείγματος χάρη, η επικύρωση. Η επικύρωση θα πάρει χρόνο. Εμείς θέλουμε πληροφορίες ε, από σας από την Προεδρία, να μας πείτε με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε Είστε βέβαιοι ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν την πολιτική βούληση να ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωση πριν το τέλο του έτου, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε και τα χρήματα, το, το ταμείο. Διότι εφόσον πρόκειται για ένα πακέτο, το ΠΔΠ δεν μπορεί να προχωρήσει χωρί το ταμείο και το ταμείο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρί το ΠΔΠ. Εφόσον θεωρούμε ότι είναι πακέτο, έτσι. Είναι συμπληρωματικέ οι πολιτικέ. Οπότε εμεί βεβαίω είμαστε ε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είμαστε ε, προετοιμασμένοι, έχουμε την εντολή μα. Στην πρώτη συνάντηση παρουσιάσαμε την εντολή μα στη Γερμανική Προεδρία. Ελπίζουμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση να έχουμε και κάποια απάντηση από τη Γερμανική Προεδρία ε, για λογαριασμό του Συμβουλίου. Ποια είναι η αντίδραση στην πρότασή μας για το πι Ευχαριστώ η Μαγκρίντα Μάρκε τώρα από του S&D, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε ο κ. Σάλμπρεχτ για το χρονοδιάγραμμα. Όντω, μα ενδιαφέρει ιδιαίτερα να φτάσουμε σε συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι σαφές και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού στα τέλη Ιουλίου. Εκεί λέμε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία στα τέλη του Οκτώβρη θα πρέπει να περάσουμε στο Plan B όπως αυτό αναφέρεται στο ψήφισμα. Δηλαδή συμφωνούμε για το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, εδώ δεν, δεν έχουμε μια συνάντηση διαπραγμάτευσης, έχουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκά Θέματα. Ε, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ε, βεβαίως, ε, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εξού και το νόημα αυτής της ανταλλαγής απόψεων με σας εδώ σήμερα. Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο σημεία. Το πρώτο έχει να κάνει με το κράτος δικαίου. Γνωρίζω ότι ο κύριος Υπουργός ε, ήταν ένας ακτιβιστής ουσιαστικά, υπερασπιστής του κράτους δικαίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Και όντως αντιμετωπίζουμε μία περίπλοκη κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχει η βούληση, η θέληση να σεβαστούμε προφανώς τις ευρωπαϊκές αξίες. Υπάρχει μια νομοθετική πρόταση επιτάπητος για το κράτος δικαίου, μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα συζητηθεί σε συναπόφαση και θα αποφασιστεί κατά πλειοψηφία και ταυτόχρονα τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να επικυρώσουν τους ιδίους πόρους για να μπορέσουμε να έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Εάν η Ουγγαρία ακολουθήσει μια τακτική πίεσης για το θέμα του κράτους δικαίου, λέγοντας ότι το Ουγγρικό Κοινοβούλιο δεν θα επικυρώσει τη συμφωνία για τους ιδίους πόρους, και μπλοκάρει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η στρατηγική της Προεδρίας στην περίπτωση αυτή. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα ζητήματα κράτους δικαίου αφενός, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι και τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών θα προωθήσουν ε, τις ευρωπαϊκές αξίες ε, και όχι άλλες Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική της Προεδρίας έτσι ώστε αυτά τα δύο εργαλεία να τα έχουμε στα χέρια μας ταυτόχρονα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα προγράμματα, όπως γνωρίζετε υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πρόταση, στα στοιχεία ε, του Συμβουλίου και τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα αριθμητικά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η στρατηγική από πλευράς Προεδρίας ποιες είναι οι προθέσεις της, έτσι ώστε να γίνουν κάποια βήματα για να δημιουργήσουμε συνθήκες επίτευξης συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες έχει το λόγο για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό. Το Κοινοβούλιο πάντα είναι υπεύθυνο και φιλόδοξο. Ουδέποτε θελήσαμε να ε, δίνουμε τελεσίγραφα ή να φέρνουμε τους υπόλοιπους ως ομήρους. Ψηφίσαμε τον ε, Αύγουστο για να ξεκινήσουμε σήμερα τις διαβουλεύσεις για τους ιδίους πόρους τον Σεπτέμβριο στην Σύνοδο Λομέλειας, θα ψηφίσουμε μια άλλη, την δική μας απόφαση. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να προχωρήσουμε γοργά γιατί χρειαζόμαστε ε, ένα πρόγραμμα ε, ανάκαμψης ε, το πρόγραμμα ανάκαμψης και αυτό θα δώσει και στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να λάβει τις αποφάσεις του και να ξεκινήσει τη διαδικασία για τις διαδικασίες κύρωσης από τα κράτη-μέλη. Μια διαδικασία που είναι απαραίτητη. Θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Πότε σκοπεύει το Συμβούλιο να ξεκινήσει και να περάσει στην κύρωση. Γιατί θεωρώ ότι είναι και λογικό, αλλά και τα θέματα είναι όχι απλώς αλληλένδετα, αλλά απαιτείται και ταχύτητα τώρα το ζήτημα των ιδίων πόρων και οι διαδικασίες των κυρώσεων θα πάρουν χρόνο. Οι διαδικασίες αυτές είναι αλληλένδετες και εμείς τις ε, διαχωρίσαμε. Σκεφτείτε να είχε κάνει το εξής το Κοινοβούλιο. Να είχε δώσει συνένεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά την κύρωση από όλα τα κρατημέλη, διότι Υπάρχει ο κίνδυνος, παρόλο που θα ήθελα να τον θεωρώ ελάχιστο, υπάρχει ο κίνδυνος κάποιο κράτος μέλος να μην συμφωνήσει, να μην περάσει σε κύρωση. Και τότε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα μπορεί να γίνει παραδεκτό, διότι δεν θα αποτελεί πλέον πακέτο. Ε, το ερώτημά μου λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ εύστοχο. Πότε θα ξεκινήσετε τη διαδικασία κύρωση, πότε θα δώσετε τη δυνατότητα να ξεκινήσουν οι κυρώσει από τα επιμέρου κράτη-μέλη. Διότι για μα ε, επήγει η επίλυση αυτού του ζητήματο. Και το άλλο ερώτημα είναι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι κανεί από εμά δεν θα κατάφερε να πείσει του συμπολίτε του ότι ένα ε, εθνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να έχει ε, δικαίωμα να επηρεάσει ένα μεγάλο ποσό που θα ενταχθεί στον προπολογισμό ε, και θα έχει μεγάλη επιρροή στην δημοσιονομική ζωή αυτού του κράτους. 380 δις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανάκαμψης. Είναι πολύ επικίνδυνο να μην μπορεί ένα κοινοβούλιο να τοποθετηθεί σε σχέση με ένα τόσο μεγάλο ποσό. Και σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική αρχή, το Κοινοβούλιο δηλαδή και το Συμβούλιο μαζί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ρόλο να διαδραματίσουν εδώ. Η Δημοσιονομική λοιπόν αρχή κάθε χρόνο στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας πρέπει να αποφαίνεται για, τα, για τις δαπάνες και τα έσοδα, για αυτά που πρέπει να καταγραφούν στον προπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει ο δημοσιονομικός κανονισμός και στη διαθεσμική συμφωνία να ενταχθούν και αυτά. Νομίζω ότι είναι απλό. Η ερώτησή μου είναι εάν να συμμερίζεστε αυτήν την ανησυχία του Κοινοβουλίου και υπέρ των πολιτών στην ουσία. Για να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και να υπάρχει και διαφάνεια αλλά και η σωστή προβολή του θέματος ώστε να φαίνεται πώς οι συνεισφορές και οι φόροι των πολιτών θα πιάνουν τόπο. Ευχαριστούμε η Βαλερή Αγέ από τους Ρινιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε Υπουργέ. Η Γερμανική Προεδρία, όπως το είπατε, στι διαπραγματεύσει θα πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για να φανεί ποιο θα είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η Ένωσή μα και οι δράσει μα. Αυτό που διακυδεύεται τώρα δεν είναι η Ευρώπη το 2021, αλλά είναι το 2028 και το 2058. Ναι, ε, εμεί στο Ευρωκοινοβούλιο και εγώ προσωπικώ πιστεύω στην Προεδρία σα, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω ότι μπορείτε να είστε ένα καλό εταίρο ε, ε, για μα και για να προχωρήσει η Ευρώπη. Δύο ερωτήσει λοιπόν για το θέμα αυτό, για του ιδίου πόρου. Δεν ξέρω ποια συγκεκριμένη έκθεση έκφραση χρησιμοποίησατε πλέον, αλλά αν, τα αν το θυμάμαι καλά, είπατε ότι με τη συμφωνία του Συμβουλίου είχαμε μια ριζική αλλαγή στο σύστημα των ιδίων πόρων. Ε, αυτό θα μπορούσε να το πει κανείς ριζικό, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία για να βρεθούμε σε μια φάση πραγματικά ιστορική σημασία και που να είναι ριζοσπαστική η αλλαγή. Εμεί στο Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε μια τέτοια ιστορική αλλαγή, διότι ξέρουμε ότι αυτά που συμφωνήθηκαν δεν είναι αρκετά. Θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα πιο ε, πιεστικό, πιο γρήγορο και δεσμεύσει. Δεσμεύσει για την υλοποίηση του συστήματο των ίδιων πόρων. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ρωτήσω για την αναφορά σας ε, ως προς την χρήση των πόρων και την αποπληρωμή των ε, δανείων, διότι αυτό ε, διαγράφτηκε από το κείμενο του Κορεπέρ, ενώ υπήρχε στο κείμενο που πρότεινε η Γερμανική Προεδρία ε, και για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μας το εξηγείτε αυτό. Γιατί συνέβη. Γιατί το Συμβούλιο πήρε απόσταση από τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν δώσει οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων. Και δεύτερο, αντιδρώντας στα λόγια σας και κάτι που το έθιξε και ο Ζωζέ Μανουέλ, ε, και σας ρώτησα γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο σε ό,τι αφορά την απόφαση για τους ιδίους ε, πόρους καταλαβαίνει πως ε, πήγε το θέμα και ότι πρέπει να κινηθούμε τάχιστα για να ξεκινήσουν διαδικασίε διαδικασίες κύρωσης. Η άποψη όμως που μας απασχόλησε και στην οποία κινηθήκαμε για το σύστημα των ιδίων πόρων εγκρίθηκε στην Επιτροπή Προπολογισμών με ευρύτατη πλειοψηφία και θα την εγκρίνουμε και στη Σύνοδο Ολομέλειας πολύ σύντομα. Ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο θα ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης, θα δώσει το πράσινο φως για την ε, κύρωση του συστήματος ιδίων πόρων από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό θέλουμε να προχωρήσει. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει ταχύτητα και το καλοκαίρι. Εργαστήκαμε, όπως είπε ο Ζωζέ Μανουέλ, εργαστήκαμε για να πάμε στο δυνατόν πιο γρήγορα και επειδή υπήρχαν και προθεσμίες που και εμείς έπρεπε να σεβαστούμε πάση θυσία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για την έγκριση τη απόφαση του ιδίου πόρου στη χώρα σα, στη Γερμανία. Μπορείτε να μα πείτε εάν προβλέπετε ήδη κάποια ημερομηνία. Έχει αποφασιστεί από την Ομοσπονδιακή Βουλή, από το Bundestag, μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίε κυρώσεων και τα κοινοβούλια της Γερμανίας θα κυρώσουν τάχιστα ακόμη και πριν υπάρξει η κοινή συμφωνία με το κοινοβούλιο για τα θέματα του CFP. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Άντρεσεν για τους πρασίνους. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μαζί σας και πραγματικά ε, και εμείς ευχόμαστε να προχωρήσουμε. Το Κοινοβούλιο δεν θέλει καθόλου να υπάρξει αδιέξοδο στην όλη διαδικασία. Θέλουμε μια καλή λύση τις επόμενες εβδομάδες και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Παρόλα αυτά, άποψή μας, άποψη του Ευρωκοινοβουλίου είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη μεταβατική περίοδο, γιατί αυτή, αυτό το γεφύρωμα που θέλαμε, αυτό το λεγόμενο bridge, δεν υπήρξε στο τελικό πακέτο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τις κατάλληλες δημοσιονομικές αποφάσεις που να μας φέρουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι όταν οι καταστάσεις είναι πολύ περίπλοκες, Έχουμε προβλήματα με τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνολικά. Στην απόφαση του Κοινοβουλίου πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε ταχθεί κατά των ε, περικοπών που πρότεινε το Συμβούλιο κατά 9,3 δισεκατομμύρια, 7,6 δισεκατομμύριο ε, για την κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, 17 ε, δισεκατομμύρια για το Ταμείο Δικής Μετάβασης, εδώ χρειάστηκε να αγωνιστούμε. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, δεν εκπροσωπούμε απλώς την ε, άποψη του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα ερχόμενα χρόνια, και κάτι το οποίο είχαμε αναλάβει από κοινού ευθύνη. Το βρίσκω λοιπόν λίγο περίεργο που ακούστηκαν στα γερμανικά μίντια απόψει από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πρόσφατα ότι το Κοινοβούλιο έχει δυσκολέψει τα πράγματα. Ε, δεν είναι προσπάθεια να δυσκολέψουμε τα πράγματα, το να ζητάμε περισσότερα για τα πολύ σημαντικά προγράμματα. Δεν με ε, κάνει απλώ να αισθάνομαι λοιπόν άβολα, αλλά με ενοχλεί κιόλα κάτι τέτοιο. Οι αριθμοί που έχετε προτείνει ω Συμβούλιο ε, πολύ σοβαρά μα απασχόλησαν. Δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί προτάθηκαν και για τα συγκεκριμένα προγράμματα όταν θέσαμε ερωτήσεις δεν λάβαμε απάντηση για τις περικοπές. Ε, Ίσως υπάρχουν αντιρρήσεις από το ένα ή το άλλο κάτω μέλος, αλλά περιμένουμε από εσά ή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, τέλος πάντων από την Προεδρία του Συμβουλίου, για αυτές τις πτυχές να, ε, τοποθετείτε, να τοποθετηθείτε κάπως. Διότι τις ερχόμενες εβδομάδες θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για ριζικές αλλαγές και θα χρειαστεί να συμφωνήσουμε. Φυσικά και πρέπει να περάσουμε σε συμβαστικές λύσεις, αλλά θέλουμε και ταχύτητα. Εύχομαι λοιπόν αυτά να τακτοποιηθούν στο πλαίσιο της Προεδρίας τις ερχόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ να περάσω στους συζητητές τώρα. Πρώτα για το πι δελτα πι, ο κύριος Κιόλνεφ έχει το λόγο για το Renew. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ Ρότ που ε, συζητάτε σήμερα μαζί μας έστω ε, και ψηφιακά για αυτό το ζήτημα. Πραγματικά είναι ε, θετικό το γεγονός ότι γίνεται μια συζήτηση με την Προεδρία του Συμβουλίου. Μα είπατε ότι είναι σημαντικό να φτάσουμε γρήγορα σε μια συμφωνία και αυτό είναι σημαντικό για μα. Εμεί εδώ και δύο χρόνια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένουμε τι διαπραγματεύσει. Η δική μα δηλαδή η θέση ήταν ανέκαθεν γνωστή και ξεκάθαρη. Επιτέλου βλέπουμε τώρα να είναι και σαφή η θέση του Συμβουλίου Οπότε να πούμε εδώ ότι οι πραγματικέ δυσκολίε σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις οφείλονταν ακριβώς στο Συμβούλιο και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω, εμεί θέλουμε να φτάσουμε σε μια καλή συμφωνία, όχι απλώ και μόνο σε μια οποιαδήποτε συμφωνία και προ αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να κινηθούμε. Αναφερθήκατε κι εσεί βέβαια στι πολύ δύσκολε διαπραγματεύσει ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και που διάρκησαν και το Σαββατοκύριακο και ούτω καθεξή. Το γεγονό όμω ότι ήταν δύσκολε αυτέ τι διαπραγματεύσει, δεν σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει απλά με τα όσα συμφώνησαν τα κράτη-μέλη. Αφού μας είπατε ότι ε, δώσαμε και πολλές ε, ε, οθήσεις σε αυτή τη συζήτηση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να πούμε ότι ακόμα δεν τις έχουμε εκφράσει πλήρως. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τα επιμέρους προγράμματα δεν έχει ξεκινήσει η διαπραγματεύση. Και έρχομαι λοιπόν τώρα στο, για τα αυτά. Αναφερθήκατε για παράδειγμα στο μηχανισμό σε ό,τι αφορά ε, το κράτος δικαίου που για πρώτη φορά προβλέπετε. Αλλά ταυτόχρονα είπατε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ερμηνεία, αν θέλετε ε, αυτής της Και πράγματι θα πρέπει να διευκρινίσουμε τώρα ακριβώς το τι ε, σημαίνει εδώ. Γιατί ε, δεν ωφελεί σε τίποτα να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίο ε, τελικά δεν ε, ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο και δεν εφαρμόζεται σωστά. Ακριβώ και με το άρθρο 7 του κανονισμού το ίδιο. αυτό το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε. Και εγώ λοιπόν αναμένω και το λέω αυτό πολύ εμφαντικά και ω νέο Ευρωβουλευτή από την Προεδρία το να, να μας βοηθήσει να επιτύχουμε ακριβώς μία ε, ε, ε, μια διαπραγμάτευση και μια συμφωνία με τον τρόπο που θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέω πρώτα. Παρακαλώ σεβαστείτε το ένα λεπτό, αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέλος της συζήτηση. Ο κύριος Ζήλε για το ECR έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, thank you, chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, και τον Υπουργό που είναι μαζί μα σήμερα. Βεβαίω να γνωρίζουμε ότι είναι διαφορετικό το νομικό καθεστώ ε, για τα διάφορα αυτά πακέτα, πι ε, ταμείο ανάκαμψη ε, και βεβαίω το θέμα του κράτου δικαίου. Βεβαίω αυτά τα διαφορετικά νομικά καθεστώτα οδηγούν ότι, στο ότι βεβαίω εμεί δίνουμε μεγάλη έμφαση στο πι έχουν σχέση με τη γεωργία, έχουν σχέση με τη συνοχή, πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα θέλαμε έναν οδικό χάρτη λοιπόν ε, για το πώς βλέπετε να προχωράτε στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε να επιβραδυνθεί ε, η διαδικασία του Ταμείου Ανάκτηση, εάν έχουν προβλήματα με την επικύρωση, διότι για κάποιες χώρε ε, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία. Θέλουμε να μα πείτε λοιπόν Πού βλέπετε εσείς να υπάρχουν περιθώρια συμβασμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόκαλης τώρα για την ΚΟΕ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό και την ομάδα διαπραγμάτευση για όλη τη δουλειά που έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες. Το Κοινοβούλιο προσπαθεί να φτάσει σε μια ιστορική γρήγορη συμφωνία Θέλω να σας ρωτήσω, δεν έχουν τεθεί ήδη πολλά ερωτήματα, θέλω να σας ρωτήσω για το περιβάλλον. Χθε σε αυτό το περιβάλλον είχαμε μια παρουσίαση μιας μελέτης που δείχνει ότι το 30% για την κλιματική αλλαγή ε, έχει μετρηθεί με τρόπους ε, μη διαφανείς ε, και μη κατανοητούς για τους πολίτες τελικά. Ε, εσείς συμφωνείτε με την άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής αυτής ότι χρειαζόμαστε μια γρήγορη και αποτελεσματική αλλαγή ε, στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ σε ό,τι φορά περιβαλλοντικά ζητήματα ή θα πρέπει να περιμένουμε για αργότερα. Thank you. Now the, on uh, resources shadow... Ευχαριστώ και τώρα οι σκιώδεις συγητές ε, για, το, για τους ιδίους πόρους. Πρώτα κυρία Λαπόρτ. Όχι, κυρία Γκίζε για τους πράσινους. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank, Herr Staatsminister Ruth. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Υπουργέ Ροτ. Λέτε ότι είναι Σημαντικό εδώ να συζητήσουμε και βεβαίω σε τέτοιου τραχώδει καιρού είναι σημαντικό να μπορούμε να συζητήσουμε. Ω Γερμανίδα βεβαίω ε, μα ενδιαφέρει ε, ότι ε, σήμερα θα πρέπει και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, που δυστυχώ σήμερα δεν είναι εδώ, να αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολίτε του. Το βρίσκουμε λοιπόν λυπηρό που ε, δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο εδώ από το Υπουργείο. Θα ήθελα να μα πείτε τώρα για. αν μπορείτε να μα πείτε πιο συγκεκριμένα τι χρονοδιάγραμμα έχει υπόψη του το Συμβούλιο. Μπορείτε να μα δώσετε χειροπιαστέ πληροφορίε. Πότε θα ξεκινήσουν οι διαδικασίε, ε, γιατί έχουμε ακούσει από τον Επίτροπο Τζεντιλόνι, για παράδειγμα, ότι ο ψηφιακό ε, φόρος, ο φόρος για τις ψηφιακές εταιρείε, μπορεί να ξεκινήσει φέτος, μπορεί και όχι, έχουμε ακούσει από αλλού. Θα πρέπει λοιπόν να μας πείτε κάτι περισσότερο για το πρόγραμμα. Και μια σύντομη ερώτηση, μια δεύτερη ερώτηση, κάτι που δεν έχει ακόμα φυγεί στο Συμβούλιο, αλλά ίσως υπάρχει δυνατότητα να, ε, να προταθεί κάτι καλύτερο στο Συμβούλιο, είναι για το gender mainstreaming, την ευθυγράμμιση των διδυστριάστες του ρόλου των φύλων και τις σχετικές πτυχές εδώ, ε, ξέρετε ότι αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και για τους άντρες αλλά και για τις γυναίκες, ε, όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας λοιπόν, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόκειται να ασχοληθεί με αυτό και τι θα κάνει η Γερμανική Προεδρία για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στου υπόλοιπου συναδέλφου. Κάτσε Κατστιάη, παρακαλώ να σεβαστείτε το μονόλεπτό σα. Αν θέλετε να προλάβουμε να ακούσουμε και τι απαντήσει του Γερμανού Υπουργού. Πρώτα απ' όλα ο κύριο Κολακούσιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Κύριε Υπουργέ, βρισκόμαστε στην πιο βαθιά κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών τα τελευταία 15 χρόνια. Τα τελευταία 50 χρόνια. Εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν στην ανεργία, εκατομμύρια χιλιάδες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση και ένας από τους τρόπους αυτούς είναι να χρησιμοποιήσουμε τους ιδίους πόρους και να φορολογήσουμε τις χρηματοπιστωτικές ε, διαδικασίες ε, τις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνίας που αυτή τη στιγμή κερδίζουν, έχουν κέρδη από την κατάσταση αυτή. Ένας άλλος τρόπος είναι να χρεωθούμε. Αυτό όμως σημαίνει ότι η μελλοντική γενιά θα, θα, πρέπει να πληρώσει αυτό το χρέος. Το πλεονέκτημα αυτών των ιδίων πόρων είναι ότι φορολογούμε αυτούς που έχουν τα κέρδη τώρα, αυτούς που κερδοφορούν τώρα. Εγώ χαίρομαι που η Γερμανία προεδρεύει του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή, διότι μας έχετε δείξει ότι ξέρετε πώς να διαχειρίζεστε ορθολογικά τον προϋπολογισμό. Ξέρετε πώς να δαπανείτε τα χρήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω περισσότερα από αυτού. He's not there. Mr. Kous, ID. Ο κύριος Κούς για την ID. Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ εγώ διαρωτώ γιατί δεν γίνεται λόγος ε, για το συνολικό κονδύλι αυτού του πακέτου. Ε, δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται εδώ. Στην, στον τύπο αναφέρεται ένα δισεκατομμύριο ακόμα και 74 εκατομμύρια κάτι τέτοιο γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Μήπω, επειδή δεν έχουν γίνει σχετικοί υπολογισμοί με βάση το ΑΕΠ, ισχύει το 1%, ισχύει το 1,07% όπως αξιώνει το Συμβούλιο, 1,11% με βάση την, ε, τα όσα θέλει η Επιτροπή, 1,3% με βάση τα όσα αναφέρει το, ε, ε, αξιώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μετά το 10% που αναφέρθηκε ε, και τη μείωση ε, λόγω του COVID. Όλα αυτά λοιπόν δεν μου απαντώνται, δεν υπάρχουν διευκρινήσεις. Και επίση διαρωτώ με για παράδειγμα, αν υπάρξει μελλοντικά ανάκαμψη τη οικονομία, θα υπάρξουν και ανάλογε αναπροσαρμογέ. Τι ακριβώ έχει προβλεφθεί. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα για τις νομοθετικές διαδικασίες να μου πείτε ε, εάν ε, τα διάφορα προβλήματα που, που υπάρχουν αν πιστεύετε ότι θα έχουν ε, επιληθεί ως το τέλος της χρονιάς. Γιατί υπάρχουν διαδικασίες στο Κοινοβούλιο και διαδικασίες κύρωσης στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, αγορά κεφαλαίων θα πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες και να έχουν μάλιστα ξεκινήσει και πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης. Ευχαριστούμε κύριο Λεαροτερίου ε, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για αυτήν την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Κύριε αγαπητέ Μιχαήλ, ήμασταν μαζί στο περασμένο Δεκέμβριο στο Βερολίνο όπου λέγατε ότι θα χρειαστεί ένα μεγάλο πακέτο ιδίων πόρων και λέγατε μπροστά σε όλους ότι καλή η φορολόγηση του πλαστικού αλλά είναι μόλις 5 δις και θα μειωθεί. Χρειαζόμαστε τη φορολόγηση του πλαστικού, αλλά δεν φτάνει. Το είπε και η Βαλερία αυτό. Ποια είναι λοιπόν η λύση για να έχουμε ένα πιο σημαντικό, ένα πιο βιώσιμο σχέδιο και ποια είναι η λύση για να σιωπήσουν όσοι λένε ότι το σχέδιο αυτό ανάκαμψη θα μας κοστίσει πολλά χρήματα. Κάποιοι το λένε στη Γαλλία, στη Γερμανία θα μας κοστίσει πολύ αυτό το σχέδιο, αυτό το ταμείο. Πώς μπορούμε να έχουμε λοιπόν βιώσιμες βιώσιμη χρηματοδότηση για το Green Deal. Ήδη το 2012 ω βουλευτή ήσασταν υπέρ τη ε, φορολόγηση των ε, χρηματοπιστικών συναλλαγών. Ω υπουργό αργότερα το 2015 λέγατε ότι ήρθε η ώρα να πάρει μια απόφαση η Ευρώπη για να φορολογηθεί η χρηματοπιστωτική συναλλαγή. Το είπε και η, Γερμα... η κυρία Μέρκελ ω προτεραιότητα τη Γερμανική Προεδρία. Είναι και δική μα προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε μια πραγματική φορολόγηση των ε, χρηματοπιστικών συναλλαγών από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Έτσι θα μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε όλα αυτά τα χρήματα που χρωστάμε και να έχουμε και χρήματα για την απασχόληση, για την υγεία, για την έρευνα, για το Green Deal. Εάν είναι προτεραιότητα λοιπόν τη Γερμανική Προεδρία ε, ξέρουμε ότι μπορούν να λυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα. Από το Σεπτέμβριο του 2011 η οδηγία είναι επιτάπητο. Δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα. Είπατε ότι θέλετε να δουλέψετε μέρα-νύχτα για να φτάσουμε σε συμφωνία. Το Κοινοβούλιο συμφωνεί να φτάσουμε σε συμφωνία, να δουλέψουμε μέρα-νύχτα για να έχουμε μια πιο σημαντική χρηματοδότηση για το πει. Ποια είναι η χρηματοδότηση για να εργαστούμε μέρα-νύχτα για μια φιλόδοξη ε, συμφωνία. Madame Keller. Merci beaucoup, euh, η κυρία Κελέρ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να υποστηρίξω τα ερωτήματα της ε, δημοκρατικής ομάδας, ιδιαίτερα ε, αυτά που τέθηκαν για τους δύο σπόρους και τον ε, απαραίτητο χαρακτήρα τους, την ισορροπία στο σχέδιο, ε, οι προθεσμίες επικύρωσης, ιδιαίτερα οι γερμανικές προθεσμίες και βεβαίως το θέμα ε, των, της συμμόρφωσης και των διαφόρων όρων. Θέλω όμως να θέσω ένα άλλο ερώτημα όχι για ένα οικονομικό ζήτημα, αλλά για την υγειονομική κρίση. Η Γερμανική Προεδρία, την οποία εκπροσωπείται εδώ σήμερα το απόγευμα, κάνει μια προσπάθεια εναρμόνισης ό,τι αφορά τα υγειονομικά κριτήρια, τα κριτήρια ανάλυσης πρώτα απ' όλα, αλλά και εφαρμογής της προστασίας από την ε, εξάπλωση της πανδημίας. Εσείς ε, είστε επικεφαλής του συντονισμού. Εδώ και κάποιες ημέρες βλέπουμε ότι η Ευρώπη είναι απούσα σε αυτήν την κοινή διαχείριση της ε, υγειονομικής κρίσης. Ευχαριστώ κυρία Κέλλερ. Ο κύριος Χόινσικ έχει το λόγο. Δεν είναι εδώ. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Υπουργό. Λοιπόν, κύριε Ροτ, έχετε το λόγο. Ήταν πολλά τα ερωτήματα και τα σχόλια που ακούστηκαν. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, βουλευτέ, σα ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας για την κριτική που ασκήσατε και να πω εισαγωγικά το εξή. Κανέναν δεν εκβιάζουμε και σε κανέναν δεν ασκούμε αθέμητες πιέσεις. Εσείς ασκείτε το ρόλο σας ως Κοινοβούλιο και για μία ακόμα φορά το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούνται να διαπραγματευτούν. Και όπω σε κάθε ζωντανή κοινοβουλευτική δημοκρατία, θα πρέπει να γίνουν σκληρέ διαπραγματεύσει ανάμεσα στα όργανα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο τέλο σε συμβιβασμού. Και έχω την εντύπωση, αξιότιμη κυρίε και κύριοι ε, βουλευτέ, ότι έχουμε προσεγγίσει αρκετά τις απόψεις μας αμοιβαία ε, και βέβαια παραμένουν κάποια ακόμα εκκρεμή σημεία ε, στα οποία οι απόψεις μας ε, εξακολουθούν να διαφέρουν. Και υπάρχει βέβαια και μία διαφορά ε, εδώ σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς λήψη αποφάσεων μεταξύ των δύο οργάνων. Εσείς αποφασίζετε με πλειοψηφία και εμεί ε, στο Συμβούλιο αποφασίζουμε με ομοφωνία. Ε, και νομίζω πως εύκολα μπορείς να καταλάβει πόσο δύσκολο ήταν να φτάσουμε στο, στο επίπεδο φιλοδοξίας αυτό που φτάσαμε. Και νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε και σε έναν βαθμό περήφανοι γι' αυτό. Γιατί πραγματικά, αν παραμείνουν από κοινού ω πακέτο δηλαδή προ διαπραγμάτευση το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και το Next Generation EU, ε, τότε έχουμε φτάσει σε ένα συνολικό πακέτο το οποίο υπερβαίνει σε μεγάλο βαθμό τι προσδοκίε όλων των όργανων. Και από εκεί και μετά έχουμε προβλέψει πολλά και σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την έρευνα και το, την κλιματική αλλαγή. Και εδώ μπορείτε να, να αναφέρετε τα όσα λέω εγώ, τα όσα λένε και άλλοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Ε, μπορείτε προφανώς να αναφέρετε τα όσα, το ότι επιθυμούσαν διάφοροι περισσότερα, αλλά τελικά έχουμε φτάσει σε ένα συμβιβασμό, ο οποίος, όπως ανέφερα ήδη, χρειάστηκε τις υποχωρήσεις και την ε, γαλακτικά από την πλευρά όλων. Και σε ό,τι αφορά ε, της, ε, την έλλειψη περιθωρίων, αν θέλετε, για μεγάλες ε, αλλαγές σε ό,τι αφορά τα όσα θέλουμε να προβλέψουμε, πράγματι υπάρχουν, βρισκόμαστε σε μια, μια πολύ σημαντική κρίση, η οποία βέβαια δημιουργεί περιορισμού σε ό,τι αφορά τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και αυτό γιατί με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χάσαμε ένα κράτος μέλος ε, ε, του οποίου η συνεισφορά και η συμμετοχή στον προπολογισμό ήταν σημαντική και θα πουσιάσουν αυτά τα κονδύλια ε, στο μέλλον. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν περισσότερο, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και βέβαια δεν λέω ότι κάτι τέτοιο είναι λάθο. Απλώ λέω ότι οι προϋποθέσεις πλέον ήταν διαφορετικές και σε σχέση με την κρίση και σε σχέση ε, με το Brexit, σε σχέση με το τελευταίο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Από εκεί και μετά, ε, θεωρώ σε ό,τι αφορά το mainstreaming της ε, κλιματικής αλλαγής ε, πραγματικά θεωρώ πως ε, θέτουμε εδώ πραγματικά ένα ε, είμαστε υποδειγματικοί σε ό,τι αφορά το 30% των μέσων και 40% αν βάλουμε και την ε, τη γεωργική πολιτική. Άρα λοιπόν πράγματι σε σχέση με το mainstreaming θα πρέπει πράγματι να εξασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται για αφηρημένε δεσμεύσει, αν θέλετε, γενικόλογε, αλλά πραγματικά για πολύ συγκεκριμένε δεσμεύσει. Και θα πρέπει πράγματι εδώ να έχουμε υψηλό βαθμό δέσμευση, δεσμευτικότητα. Εγώ δηλαδή ε, από κοινού με την ε, Σουηδό ομόλογο μου είχαμε επιμείνει πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το mainstreaming τη κλιματική αλλαγή και προ, προφανώς μπορείτε να αναμένετε ότι εγώ θα βρίσκομαι στο πλευρό σας σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή ε, θα πρέπει αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, πολιτές δηλαδή δημοσιονομικό πλαίσιο από κοινού με τον Next Generation EU, να οδηγήσουν και στο κατάλληλο mainstreaming προκειμένου να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Και πραγματικά θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια καλή κοινή λύση. Και έρχομαι τώρα στην ε, απόφαση ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους. Εντάξει, δεν μου αρέσουν πάντοτε έτσι ιστορικές, αν θέλετε, ε, και βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά πραγματικά εγώ δεν θα μπορούσα, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, η προσωπική μου άποψη όταν αφορά τους ίδιους πόλους ένωσης, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πριν από κάποιους μήνες ότι θα ήμασταν σε θέση να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα ομόφωνα. Ούτε καν με ειδική πλειοψηφία δεν μπορούσαμε να φανταστώ ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν εδώ υπήρξε πραγματικά, επιτύχαμε μία ρίζοσπαστική αν θέλετε, μία εκτεμελίων αλλαγή σε ό,τι αφορά του ίδιου ε, πόρου. Ε. Και βέβαια, ναι, έχουμε ένα πρώτο βήμα εδώ σε ό,τι αφορά την, ε, τον φόρο κατά πλαστικά. Υπήρξαν και περαιτέρω προτάσεις που έθεσαν, έθεσε το Κοινοβούλιο και εξακολουθούν να εξετάζονται. Αλλά από εδώ και ε, πέρα τώρα θέλουμε πιο συγκεκριμένες προτάσει και ε, αναμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα συγκεκριμένο χάρτη πορεία, ένα roadmap για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σχέση με αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Και αυτό που θέλετε και εσεί βέβαια, να υπάρξει δηλαδή κάτι πιο συγκεκριμένο. Όμως ε, παραμένει γεγονός ότι ε, το ζήτημα των ιδίων πόρων αποτελεί ένα ιδιαίτερα λεπτό, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Αναφέρθηκε πριν από ε, λίγο ότι τα έσοδα από τους νέους ίδιους πόρους από το 2020 και μετά θα χρησιμοποιηθούν για την εξάλληση αν θέλετε της, των, οδοτήσεων. Οπότε, ε, πραγματικά η λογική εδώ είναι απλή. Ε, δύο ε, τρόποι υπάρχουν να πληρώσουμε τα δάνεια μας. Ή τα κράτη-μέλη ανταποκρίνονται σε αυτές τις ενισχύσεις ή ζητούμε συμπληρωματικούς ίδιους πόρους. Αυτά είναι τα δύο εργαλεία, αν θέλετε, δύο τρόποι, αν θέλετε, για να εξοφλήσουμε τα, τα δάνεια αυτά. Άρα λοιπόν, νομίζω πως είναι αυτός ο σωστός τρόπος να, και, έχουμε επιτύχει μια σωστή λύση. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα του governance, τη διακυβέρνηση, νομίζω πως και εδώ έχουμε ε, ε, κοινή άποψη. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε εδώ μια, με μια πολύ σημαντική απόφαση σε ό,τι αφορά ακριβώς και την ενσωμάτωση του Next Generation EU μέσα στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να αναλάβουν και τις ε, αντίστοιχες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις ως συνομοθέτες και για τα ζητήματα τα δημοσιονομικά, το ε, Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε και σε σχέση με αυτό το ζήτημα να φτάσουμε σε μια λογική, ικανοποιητική λύση η οποία θα ανταποκρίνεται με καλύτερο τρόπο ακριβώ τι αρμοδιότητε ω συνομοθέτε του ε, Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ρεσιμότητε, προποθέσει δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη Κυρίε του κράτους δικαίου. Ε, πολλοί από εσά ε, με γνωρίζετε και από το παρελθόν. Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ε, πραγματικά πρόκειται για ένα ζήτημα που και εσύ, Μαργαρίτα, ε, έχει προωθήσει σε μεγάλο βαθμό και στο παρελθόν, αλλά εδώ ε, δεν έχουμε να κάνουμε με την άποψη τη δική μου ή την άποψη της κυβέρνησης της Γερμανίας έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα σημαντικό βήμα το οποίο καλείται να ε, κατάφερε να κάνει ουσιαστικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Συμβούλιο. Αυτό όμως που δεν θα δεχτώ ε, είναι να υπάρχει ένα, ένα δίλημα, αν θέλετε, τη τάξη του είτε κονδύλια, είτε χρήματα, είτε κράτο δικαίου. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει. Δηλαδή ένα τέτοιο αφήγημα, αν θέλετε, δεν θα πρέπει να το ασπαστούμε εμεί. Έγινε μία πρόταση η οποία αποτελεί μια μεγάλη υπέρβαση, αποτελεί κάτι το καινοτόμο ε, και θα διαπραγματευτούμε πλέον αυτή την πρόταση επί ίσης όρης με εσάς ως συνομοθέτη. Με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρούμε πως με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ε, γίνει και η σωστή ε, περικοπή που χρειάζεται το κοντιλίο. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το σημαντικότερο θέμα. Ε, τέθηκαν ερωτήματα σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα πότε για παράδειγμα κάτω βουλή της ε, Γερμανίας θα εγκρίνει την απόφαση ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους και ούτω καθεξής. Επαναλαμβάνω λοιπόν για μία ακόμα φορά το, ε, τη δική μου παράκληση να αξιολογήσετε από τη δική σας ε, πλευρά το κατά πόσο αυτή η συνολική δέσμη προτάσεων που αποτελείται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Next Generation EU και το κράτος δικαίου, κατά πόσο λοιπόν θα είχε νόημα να διασπάσουμε αυτό το πακέτο θεωρώ πως αυτή η ισχύ, αν θέλετε, αυτού του πακέτου είναι το γεγονό ότι συγκεντρώνει διαφορετικά συμφέροντα και εξυπηρετεί διαφορετικά συμφέροντα από διαφορετικού τομεί. Υπάρχουν δηλαδή κάποια κράτη-μέλη τα οποία σε τεράστιο βαθμό από το πολιτέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Άλλα κράτη-μέλη τα οποία έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση αναμένουν ε, ε, υποστήριξη σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ε, πανδημίας. Ενώ υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη τα οποία θα υποφεληθούν ιδιαίτερα από τις ε, ρυθμότητε σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν θέλουμε να διασπαστεί αυτή η δέσμη προτάσεων, αυτό το πακέτο. Γιατί τελικά προς το συμφέρον όλων θα είναι το να καταλήξουμε σε μια συνολική αλλά και ταχεία λύση. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι πολύ επικριτικός απέναντι ε, σε αυτήν την αναφορά που γίνεται σε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ε, που ουσιαστικά θα επιμήκυνε το, το status quo. Ε, κάτι τέτοιο δεν θα μας ε, επέτρεπε να εξυγχρονιστούμε, να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι ανάμεσα στο, απέναντι στο μέλλον, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά και το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν, η συμφωνία που θα φτάσουν σε ό,τι αφορά το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο των Next Generation e και το κράτος δικαίου θα αποτελέσει την βάση για ή αν θέλετε τον εναρκτήριο λάκτισμα για να ξεκινήσει η συμφωνία στα, στο επίπεδο των επιμέρους κρατών μελών σε ό,τι αφορά τους ίδιους πόρους. Και με βάση τα όσα ε, ακούω υπάρχει μεγάλη ε, ε, θέληση, βούληση πολιτική και για παράδειγμα στη δική μου ε, χώρα ε, ως προς το ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Και αυτό είναι και το αίτημα που ακούμε και γενικά από τους πολίτες, ότι θα πρέπει δηλαδή τα μέτρα αυτά να ληφθούν και να εφαρμοστούν άμεσα. Ταχύτατα. Και εγώ βέβαια από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ. Οπότε σας παρακαλώ για μία ακόμα φορά. Ε, να μην διασπάσουμε αυτό το πακέτο, να παραμείνει ως πακέτο και να συζητηθεί. Και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω συζητήσεις και χωρίς βέβαια να θέλω να είμαι προκλητικός σας λέω ότι βέβαια εδώ τον, τον ε, ε, κύριο ρόλο τον έχουν αναλάβει οι Υπουργή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την ε, ε, δική μας Προεδρία του Συμβουλίου να ε, καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατό σε μια συμφωνία σε σχέση με αυτό το συνολικό πακέτο πολιτούς, δημοσιονομικού πλαισίου και Generation Ευχαριστώ ε, θερμά όλους εδώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ τον ε, ε, πρόεδρο, την Μαργαρίτα Μάρκες, τον κύριο Φερνάντες, τον Γιάνν Όλμπριχτ. Έχουμε συνειδηθεί επανειλημμένα και στο παρελθόν και νομίζω πως αυτή η συνεργασία μας που έχει βασιστεί σε εμπιστοσύνη θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί και στο μέλλον. Προφανώς θα υπάρξει διαμάχη εντό εισαγωγικών μεταξύ μας στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί σε αυτή τη διαμάχη μας προς όφελος των πολιτών μας και ας το κάνουμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστούμε Πουργερότ και ευχαριστούμε για τον ενθουσιασμό σου στο θέμα αυτό. Συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό για να φτάσουμε σε συμφωνία. Ε, είναι πολλή δουλειά που μένει να γίνει ακόμα, αλλά είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε και καυγά αν χρειαστεί, αλλά επικοδομητικά θα γίνουν όλα αυτά και με θετικό πρόσημο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. The next meeting for the people present. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 21 Σεπτεμβρίου της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.